Καλημέρα, καθίστε παρακαλώ. Χαίρομαι που σήμερα είναι η ιστορική ημερομηνία που συνεδριάζουμε με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Σας καλωσορίζω και τον Πρόεδρο Κλοντ ε, για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τη, συμφωνία, για την οδηγία PIF εισηγητής Λόπε Αγγελάρ ήταν συνεισηγητής στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. και νομίζω ότι είναι πραγματικά ιστορική ημερομηνία και δίνω το λόγο στον συνάδελφο Κλοντ Μορά. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. για να παρουσιάσω τον συνεισηγητή Λόπε Αγγιλάρ, να κάνω μια σύντομη εισαγωγή και να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Ο κύριος Αγγιλάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ τους συνεισηγητές αυτή τη δύσκολη ε, οδηγία. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και όπως είπατε είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή τη στιγμή για την οδηγία PIF όπως αποκαλείται που ε, είναι η οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την καταπολέμηση της απάτης. Ένας ε, πολύ σύνθετος φάκελος πρόκειται για ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο τονίζει ε, στον ύψιστο βαθμό τη σημασία του χώρου δικαιοσύνης και ελευθερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ευρωπαίος νομοθέτης ε, ασχολείται με το θέμα αυτό για τον τομέα της απάτης, ε, ένα θέμα που απασχολεί τα κράτη-μέλη και ο Ευρωπαίος Νομοθέτης ε, προσπαθεί να καλύψει όλους τους τομείς ε, για τους οποίους ε, υπάρχουν υποψίες, ένας τομέας που θεωρείται το εθνική κυριαρχία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε να προσθεθεί ο ΦΠΑ στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας εφόσον πρόκειται για έναν πόρο, οικονομικό πόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και διαπραγματευόμαστε πάνω από τρία χρόνια, σχεδόν τέσσερα χρόνια διαπραγματευθήκαμε την οδηγία αυτή. Πάντοτε έχοντας κατά ότι ο Ευρωπαίος εισαγγελέα θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το γραφείο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο EPPO, όπως αποκαλείται, γιατί αυτή η οδηγία, PIF, θα πρέπει να είναι υπό την αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν η δημιουργία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα για θέματα που συμπεριλαμβάνουν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, των κρατικών προμηθειών, κυρώσεις για ποινικά δικήματα και οδηγίες παραγραφής για τα αδικήματα απάτης. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το καθένα από αυτά. Καταρχήν, για, το, για την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Ένα επίμαχο θέμα, διότι εμείς θέλαμε ο ΦΠΑ να περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε την διασυνοριακή απάτη στο ΦΠΑ. Μεγάλη προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της απάτης ένα ε, ιδιαίτερα επίμαχο θέμα για τα κράτη-μέλη. Επέμειναν τα κράτη-μέλη ότι είναι αρμοδιότητα των εθνικών φορολογικών διοικήσεων. Εμείς επιμείναμε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό οικονομικό πόρο και μετά από πολλές συζητήσεις στο Συμβούλιο και σε τριμερείς διαλόγους θα συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ πάνω από το κατόφλι των 10 εκατομμυρίων ευρώ όταν ε, η απάτηση του ΦΠΑ ε, συμπεριλαμβάνει δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη. Ε, ένα κατόφλι των 3 εκατομμυρίων ευρώ είναι ήδη υψηλό και πολλές διασυνοριακές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ ξεπερνάνε τα 10 εκατομμύρια ευρώ ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στο μέλλον θα είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά. Απάτη στον τομέα των κρατικών προμηθειών. Άλλο ένα επίμαχο θέμα στο οποίο πολεμήσαμε με την κυρία Γκρέσλε και συμφωνήσαμε ότι θα συμπεριληφθεί, αλλά θα το επανεξετάσει το θέμα η Επιτροπή όταν συντάξει την έκθεση για την υλοποίηση αυτού του θέματος. Το τρίτο είναι η συζήτηση για τις ελάχιστες και μέγιστες ε, κυρώσεις. Η συμβαστική λύση περιλαμβάνει ελάχιστες και μέγιστες κυρώσεις που φτάνουν τέσσερα έτη φυλάκισης ε, για πάτες ε, άνω των 100.000 ευρώ και είναι δεσμευτικές κυρώσεις που θα πρέπει να εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη. Και τέλος η περίοδος παραγραφής Εδώ δεν θα υπάρξει απόλυτη εναρμόνιση. Μπορούμε να συμφωνήσουμε για μια ελάχιστη περίοδο 5 ετών σε όλα τα κράτη-μέλη για τα δικήματα που αναφέρονται στην οδηγία, αλλά επίσης θα επανεξεταστεί αυτή η περίοδος ε, ώστε να έχουμε τρία χρόνια σε ορισμένες περιστάσεις. Τελικά λοιπόν Μπορεί να μην έχουμε μια τέλεια συμφωνία, αλλά είναι ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός. Και παρέχει τα θεμέλια για να δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας σε θέματα ποινικού δικαίου. Στις κοινέ συνεδριάσεις των Επιτροπών ψηφίσαμε και συμφωνήσαμε για τη συμφωνία αυτή και θα πρέπει να εγκρίνουμε μία έκθεση που θα εγκρίνει την έκθεση του, το κείμενο του Συμβουλίου που συμπεριλαμβάνει τη συμφωνία των συνομοθετών, δηλαδή Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τις πολιτικές ομάδες που συμμετέσχουν στην διαμόρφωση αυτού του συμβιβασμού γιατί όλοι δούλευσαν σκληρά για να το επιτύχουμε. Και η κυρία Γκρέσλε και εγώ, συνεισηγητές, παραμένουμε, παραμένουμε στη διάθεσή σας ε, για ε, να διαμορφώσουμε περαιτέρω τις λεπτομέρειες αυτής της συμβαστικής λύσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Γκρέσλε. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ε, λάθος, λάθος δεν θα γίνει ψηφοφορία. Ο κύριος Μωράης. Ναι, η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι 6 Ιουνίου ε, και στις 15 Ιουνίου στο Στρασβούργο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Δεν υπάρχει κάτι για τα διάφορα, άρα λίγη η συνεδρίαση, η κοινή συνεδρίαση με την ΛΥΜΠΕ. Στις 15 Ιουνίου θα τα ξαναπούμε για την ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Πέρα τη συνεδριάσεως.